τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν διανεμηθεί. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις. Τα συνοπτικά πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται.